Κύριοι, αξιότιμες κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για μια ιστορική πρόκληση. Αυτή είναι που αντιμετωπίζουμε με το κύμα των προσφύγων. Χρειάζεται αλληλεγγύη και προς τα μέσα και προς τα έξω. Γι' αυτό και θα ψηφίσετε αμέσως τώρα για ένα κατεπήγον μέτρο για την μετεγκατάσταση 120.000 προσώπων που ζητούν άσυλο και που περνούν από Ελλάδα και Ουγγαρία. Η συνεχιζόμενη κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο εάν λάβουμε υπόψη την εξωτερική διάσταση του προβλήματος. Η κατάσταση στη Συρία και στις γειτονικές της χώρες επιδεινώνεται διαρκώς. Κάθε μέρα λοιπόν ξεκινούν το επικίνδυνο ταξίδι προς την Ευρώπη όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Γνωρίζουμε όλοι ότι η σύγκρουση στη Συρία βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο και δεν διαφαίνεται πολιτική λύση. Η βία έχει εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες. Χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι. Χάνουν τη δυνατότητα να παραμείνουν καν στην πατρίδα τους. Παραπάνω από τους μισούς ανθρώπους της χώρας αυτής ζουν ούτως ή άλλως σε συνθήκες υπέρτατης φτώχειας. Από 4 εκατομμύρια καταχωρισμένους Σύρους που βρίσκονται χάρη στην γενεοδορία της Ιορδανίας, του Λιβάνου και της Τουρκίας και ζουν εκεί και διαβιούν ή μάλλον θα έλεγα καλύτερα επιβιώνουν απλώς εκεί υπό δύσκολες συνθήκες και αυτό διότι οι χώρες υποδοχής, ιδίω η Ορδανία και Λίβανος, έχουν φτάσει πια στα όρια τους. Ακόμα και εκείνοι οι οποίοι προσφέρουν βοήθεια στους πιο ευάλωτους και αυτοί φτάνουν στα όρια τους. Τελειώνουν τα χρήματα του είπα του αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Πολλοί από εσά συναντήσατε τον κύριο Ρέζη τις τελευταίες μέρες. Κυρίες και κύριοι, στη μοίρα τους ανθρώπους αυτούς και ιδίω τον UNHCR. Ήδη από το Δεκέμβριο του 2014 διηρηθήθηκε οργάνωση για να εξασφαλίζει τα απαραίτητα στους πρόσφυγες επιτόπου. Η κυρία Μογκερίνη μόλις προ δύο ημερών μας υπενθύμησε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι από αυτό το ταμείο υποτίθεται ότι θα διετίθετο 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέχρι τώρα έχουν εκρέψει μόνο 41 εκατομμύρια. Από τον κοινοτικό προϋπολογισμό μόνο 5 εκατομμύρια. Τα περισσότερα μάλιστα τα έδωσαν Γερμανία και Ιταλία. Γι' αυτό παρακάλεσα τον Πρωθυπουργό κ. Μπέτελ ως Προεδρεύοντα του Συμβουλίου Υπουργών. Εφόσον βεβαίως συμφωνείτε του απέστειλα επιστολή λοιπόν αναφερόμενο στο ψήφισμά μας της προηγουμένης εβδομάδος και τον παρακαλώ, τον προσκαλώ να φροντίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση να καταβληθούν τα εκκρεμή ποσά και ζητώ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλό και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναζητήσει όλα τα διαθέσιμα κονδύλια από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για να τα διαθέσει για βοήθεια στην Ιορδανία, στον Λίβανο, όπου είναι δυνατόν στη Συρία και στην Τουρκία. Εάν δεν το καταφέρουμε αυτό κυρίες και κύριοι, τότε θα αντιμετωπίσουμε πολύ περισσότερα προβλήματα από ό,τι αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η αξιοπιστία μας εξαρτάται άλλωστε από το εάν τα χρήματα που επιθυμούμε να διαθέσουμε τις χώρες αυτές όντως θα καταβληθούν. Γι' αυτό σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας θα δημοσιεύσω άλλωστε την επιστολή. Παρακάλεσα τον Πρωθυπουργό κ. Μπέτελ ενή περιπτώσει υπάρξει έκτακτο συνέδριο, έκτακτη, έκτακτο συμβούλιο μάλλον των ε, αρχηγών κατών και κυβερνήσεων, να φροντίσει ώστε να συμφωνήσουν να διατεθούν αμέσως τα χρήματα αυτά. Κύριε Βέμπερ, εσείς. Κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε σε μια ασυνήθιστη πολιτική κατάσταση. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντικότατε προκλήσει. Γι' αυτό και υποστηρίζει η πολιτική μου ομάδα την σημερινή έκτακτη συνεδρίαση. Είναι σημαντικό το μήνυμα πρέπει να δώσουμε σήμερα ότι η Ευρώπη δηλαδή έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει τι υποσχέσει, τι δεσμεύσει τη. Θα δώσουμε σήμερα ένα μήνυμα αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Εξ ονόματο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο υποστηρίζω την θέση σα ότι πρέπει να δοθεί μήνυμα αλληλεγγύη και προ τα έξω. Το σημερινό μήνυμα είναι το πρώτο βήμα. Χρειαζόμαστε και άλλα μέτρα. Πρέπει να συζητηθούν και θέματα όπως έλεγχη των εξωτερικών συνόρων, όπως καθορισμός ασφαλών τρίτων χωρών. Όλα αυτά πρέπει να μπουν σε ένα πακέτο μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής απαντήσεως. Σήμερα, ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να δράσει. Και γι' αυτό υποστηρίζομαι τις προτάσεις σας. Ο κύριος Πιτέλα. Πολύ σύντομα, η ομάδα των σοσιαλιστών είναι απόλυτα πεπισμένη ότι σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποστείλει ένα στεναρό μήνυμα αλληλεγγύης και προσοχής προς τους πρόσφυγες, αλλά και προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Εμείς υποστηρίζουμε την επιστολή σας, συμμεριζόμαστε το πνεύμα της και το αίτημα το οποίο απευθύνεται προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο πρόεδρος Μάρτιν Σούλτ. με συγχωρείτε κύριε Πιτέλα, φαίνεται πως υπάρχει πρόβλημα με τη γερμανική μετάφραση. Θα παρακαλέσω, να τα πω στα γαλλικά, παρακαλώ την γερμανική μετάφραση. Λειτουργεί τώρα η γερμανική μετάφραση. Ωραία, ευχαριστώ κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Πιτέλα, συνεχίστε. Έλεγα κύριε Πρόεδρε ότι συμμεριζόμαστε την επιστολή σας ε, και εμείς ε, κάνουμε το αντίστοιχο αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να κινητοποιήσουν αμέσως αυτά τα κονδύλια προκειμένου να υποστηρίξουν τους πρόσφυγες στην Ιορδανία, στο Λίβανο και στην Τουρκία. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να απευθύνω εξ ονόματος όλης της μου ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δεσμεύονται αυτή τη στιγμή, αυτές τις ώρες, με πάθος, με αγάπη και πολύ μεγάλες δεξιότητες, αποδεικνύοντας την τεράστια γενεοδορία τους. Ο κύριος Thank you for the support. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ε, πρωτοβουλία αυτή. Χθε στη συζήτηση με τον κύριο Τίμερμανς ε, θέσαμε ήδη το ζήτημα αυτό, δηλαδή της έλλειψης χρηματοδότησης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης Επομένως ε, δεν μπορούμε παρά να σας υποστηρίξουμε πλήρως. Και πρέπει να σας πω ότι δεν καταλαβαίνω όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει στον προπολογισμό τη κάποια εκατομμύρια δισεκατομμύρια για να χρηματοδοτεί απευθεία ε, το Ηνωμένα Έθνη. Με τέτοια κρίση βλέπουμε να έχουν μεταφερθεί μόνο λίγα εκατομμύρια. Ελπίζω λοιπόν τώρα ε, να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε εδώ και εκεί κάποιες εξαιρέσεις. Monsieur le Président. κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να δείξουν τον ελάχιστο σεβασμό όσοι κάνουν φασαρία εδώ για τους συναδέλφους τους. Θα ήθελα και εγώ να υποστηρίξω Μην ανησυχείτε, θα μιλήσω για το διαδικαστικό και είναι το εξής το διαδικαστικό κύριε Πρόεδρε. Θα εγκρίνουμε σήμερα κατεπηγόντως ένα κείμενο. Επιμένω εξ ονόματος της ομάδος μου στο ότι εάν το Συμβούλιο τροποποιήσει ουσιοδός την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιμένω το Κοινοβούλιο ε, να ε, μπορέσει να γνωμοδοτήσει εκ νέου, γιατί έχει αυτό το δικαίωμα. Παρακαλώ, πριν νομοθετείτε, καλό είναι να ακούτε. Ευχαριστώ. <clears throat> Και πριν φωνασκείτε. Ο κύριος Φόξ. Κύριε Πρόεδρε, νωρίτερα είπατε ότι θέλετε να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη. Και ε, Ένα μετανάστη θα συμφωνούσε ίσω μαζί σα. αλλά αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη δεν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την υγεία του και έχουν τη δυνατότητα να περπατήσουν από τη Συρία στα σύνορα τη Ευρώπη. Αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη είναι στα στρατόπεδα προσφύγων στην Τουρκία και στο Λίβανο. Η ομάδα μου λοιπόν θα καταψηφίσει αυτή την πρόταση, γιατί δεν θεωρούμε ότι το να ανοίξουμε τι στήρες τη Ευρώπη σε όποιον μπορεί να φτάσει μέχρι τα σύνορα είναι η σωστή μέθοδο να του βοηθήσουμε. Και επίση θεωρούμε ότι είναι λανθασμένο για λόγου αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατάζει ή με τα δικά σα τα λόγια να υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να δεχτούν ανθρώπου στι χώρε του παρά τη θέλησή του. Ο κύριος Ηλικιώτης. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς ε, παρόλο που αυτό το ψήφισμα δεν θεωρούμε ότι είναι αρκετό, υπάρχει μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση υπάρχει πόλεμος η ευρωπαϊκή ένωση με όλους τους θεσμούς πρέπει να συμβάλλει ώστε να υπάρξει ειρήνευση στην περιοχή εν τούτης όμως θεωρούμε απαράδεκτο το ότι σήμερα κράτη μέλη κλείνουν τα σύνορα δεν βλέπουν ακριβώς αυτήν τη μεγάλη ανθρωπιστική κρίση εμείς θα στηρίξουμε αυτή την πρόταση πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις Χρειάζονται επιγόντως βοήθεια οι χιλιάδες ανθρώποι και χρειάζονται βοήθεια τα κράτη-μέλη όπως η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Ελλάδα. Γι' αυτό παρόλο το ότι ζητούμε περισσότερα, παρόλο που ζητούμε να υπάρξει μια συνολική πολιτική διαχείριση του προσφυγού, εν τούτης, ε, θα ψηφίσουμε αυτό το ψήφισμα, ε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φάραντζ. Κύριε Πρόεδρε Σούλτ, η είπατε αρμοστία για του πρόσφυγε είπε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 59 εκατομμύρια εκτοπισμένοι άνθρωποι ανά τον κόσμο. Και πραγματικά το να υπερψηφίσουμε αυτό το ψήφισμα σήμερα, αυτή την ομοθεσία, είναι σαν να αποστέλουμε μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να δεχθεί απεριόριστο αριθμό ανθρώπων. Αυτό είναι και από ε, ε πρακτική πλευρά αδύνατο. Και μήπω ήταν πιο λογικό να σκεφτούμε ε, τι λέει η Σύμβαση της Γενέβης του 1951 για τον ορισμό του πρόσφυγα. Πρόσφυγας είναι άτομο ή άτομα τα οποία λόγω της θρησκείας τους, ε, των πολιτικών πεπιθήσεων ή του προσανατολισμού τους ε, διώκονται άδικα. Αν εμεί ω κράτη-μέλη εφαρμόσουμε τη σύμβαση αυτή και θέλουμε να βοηθήσουμε του πρόσφυγε, θα πρέπει να, να έχουμε και την υποστήριξη του των πολιτών μας. Το να δεχτούμε εκατομμύρια ανθρώπους διευκολύνοντας μία έξοδο και να τη κερδοσκοπία των διακινητών και να οδηγούμε περισσότερους ανθρώπους να πνίγονται στη Μεσόγειο δεν έχει κανένα νόημα. Ο κύριος Μπορέλη, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα μου δεν έχει κοινή άποψη στο θέμα αυτό. Η Ιταλική Αντιπροσωπεία στο ιστορικό της υποστηρίζει απόλυτα το έτοιμά σας. Είμαστε πεπισμένοι Είμαστε πεπισμένοι ότι η Ευρώπη πρέπει να ε, δράσει ως Ευρώπη και τρία κράτη-μέλη δεν πρέπει να μείνουν μόνα τους να αντιμετωπίσουν αυτή την κατεπίγουσα κατάσταση. Ευχαριστώ. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας κύριε Μπορέλη και σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θεωρώ απαράδεκτη την παρέμβασή σας υπό την ιδιότητά σας ως Προέδρου εκφράζεται άποψη απέναντι στο Κοινοβουλίο. Από την άλλη μεριά δεν επιτρέψατε να γίνει συζήτηση. Εμείς συζητήσαμε να γίνει συζήτηση για το σημαντικό αυτό θέμα της ημερησίας διατάξεως και βρισκόμαστε τώρα σε μια κατάσταση ενός ιονή κοινοβουλευτισμού, ενός φαινομενικού κοινοβουλευτισμού όπου γίνεται μια δίθεν συζήτηση όπου κάποιοι που σηκώνουν το χέρι ενδεχομένως να λάβουν το λόγο και ενδεχομένως όχι βλάπτεται τον Ευρωπαϊκό Κοινοβουλευτισμό όταν σε ένα τόσο σημαντικό θέμα δεν επιτρέπεται να διεξαχθεί μια γνήσια συζήτηση. Απευθύνω έκκληση προς πάντας να διατηρήσουμε το κύρος του σώματος και σε σημαντικές αποφάσεις να επιτρέπεται η συζήτηση και όχι με αποφάσεις που λαμβάνονται στο πόδι να γίνονται δηλαδή χωρίς συζήτηση, διότι βλάπτεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η προσπάθεια κατανομής των προσφύγων που ε, αποσκοπείται με την απόφαση αυτή που λαμβάνεται με τέτοια ταχύτητα θα βρει μεγάλη αντίσταση. Χρειαζόμαστε μια λύση που να κινείται προς την κατεύθυνση να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς στην Ήπειρο όπου γεννήθηκαν και ζουν και όχι να επιβάλλουμε στις χώρες μέλη πράγματα στα οποία ούτως ή άλλως ο ευρωπαϊκός, ο ευρωπαϊκός πληθυσμός δεν συμφωνεί. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Βεχόστατ για την επισήμανση. Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κύριος Τίμερμανς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που ε, μου δίνετε το λόγο. Ο κόσμος ε, αντιμετωπίζει μια προσφυγική κρίση. Και πολύ σωστά το επισήμανε ο κύριος Φάρατς. Και θα παραμείνει για χρόνια αυτή η κρίση. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την άμεση κρίση όμως, αν θέλουμε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε και την πιο διαρθρωτική κρίση. Σήμερα ως Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουμε πολιτική πρόκληση, ανθρωπιστική πρόκληση και θα έλεγα και ηθική πρόκληση. Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε λύσεις, λύσεις που είναι ρεαλιστικές που συμμορφούνται με τις νομικές υποχρεώσεις μας, αλλά που πάνω απ' όλα συμμορφούνται και ακούν και τις, τα προστάγματα της ψυχής μας. Σήμερα, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέλω να σας πω ότι είμαστε άκρος ευγνώμονες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που κατενόησε το κατεπήγον του ζητήματος. Είμαστε ευγνώμονες στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πήρε την κατάσταση στα χέρια του και έδωσε τη δυνατότητα διεξαγωγής σήμερα της ψηφοφορίας, ούτω ώστε και τα διοθεσμικά όργανα υπό την ηγεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μπορούν να πούν στο Συμβούλιο και στα κράτη-μέλη ότι τώρα είναι η ώρα για δράση. Και αυτό βασίζεται στις ανθρωπιστικές μας αρχές. Εμείς δεν υποστηρίζουμε ότι πρέπει να ανοίξουν όλα τα σύνορα αυτό το οποίο υποστηρίζουμε είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ακούμε τη φωνή της καρδιάς μας, αυτοί οι οποίοι ε, διώκονται και οι οποίοι φεύγουν από τον πόλεμο, από τις διώξεις, είναι στις ψυχές μας, πρέπει να παραμείνουν εκεί, πρέπει να δράσουμε τώρα και ε, σας ε, ζητώ να λάβετε την πολιτική ευθύνη, να ψηφίσετε σήμερα και σας ευχαριστώ.